Colleagues, και κύριοι, καλώ ορίσατε. Παρακαλώ, καθίστε. Um, καλώ ορίσατε στην συνεδρίαση τη Επιτροπή ΣΕΝΤΕ, η οποία ακολουθείται πάρα αυτά από την κοινή συνεδρίαση τη ε, Επιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ, της επιτροπής Ασφάλεια και Άμυνας με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και έχουμε καλεσμένο το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να παρατηρήσω αυτή τη εξαρχή ότι μεταδιδόμαστε στο διαδίκτυο και σε ό,τι αφορά την διερμηνία, προτεραιότητα δίνεται στις γλώσσες των ε, μελών της ε, ΣΕΝΤΕ. Λόγω της ειδικής περίστασης έχουμε προσθέσει και άλλες γλώσσες στην Γερμανία. εγκρίνουμε αργότερα τα πρακτικά. Θα ήθελα στην παρούσα φάση να ζητήσω να εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, η σημερινή ημερήσια διάταξη και έλλειψη σχολείων και παρατηρήσεων θεωρώ ότι είναι εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη και πάρα αυτά θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στον κύριο David Μακάλιστερ. Καλώ ορίσατε, αξιότιμοι καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φωτήκα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαρά και τιμή να σας ε, καλωσορίζω στην σημερινή ε, συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την ε, Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και θα ήθελα να πω ότι είναι τεράστια τιμή και χαρά Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιέντς Στόλτονμπεργκ το ότι σα κατελωσορίζουμε στη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφαιρεώνετε το χρόνο αυτό και ήλθατε εδώ για να ανταλλάξετε απόψεις με τα μέλη των τριών επιτροπών. Είσαστε τακτικός προσκεκλημένος των επιτροπών μας και αυτό καταδεικνύει την ισχύ της δεσμευσή μας για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ αυτού του δύσκολου και χαλαπού καιρού. Νομίζω ότι πέρα από τι πολιτικέ διαφορέ που ασφαλώ έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι συμφωνούμε εν γέννη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργάζονται ακόμα πιο στενά στο μέλλον. Και οι δύο οργανώσει λοιπόν έχουν λίγο πολύ τα ίδια κράτη-μέλη και αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να βρούμε συνέργειε και τρόπου ε, συμπληρωματική δράση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε πολλά ζητήματα που μα απασχόλουν στι επιτροπέ μα τι τελευταίε εβδομάδε, πολλέ προκλήσει. και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το συνολικό πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται δραματικά του τελευταίου μήνε. και δυστυχώ ε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κρίση αστάθεια και οι συγκρούσει έχουν όλε κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο μάλλον. Και όλοι μιλάμε για την αστάθεια αυτή και τις τριβέ που επικρατούν στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δυστυχώ αυτά έχουν επιτυνωθεί. Οι εξέλιξεις στα Δυτικά Βαλκάνια μα ανησυχούν ιδιαίτερως ε. και στη Συρία και ό,τι αντίκτυπο συνεπάγεται αυτό για την σταθερότητα της ε, Μέση Ανατολή στο σύνολό τη ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και τις συνέπειες τη τρομοκρατική αυτή ιδεολογία, τη τρομακτική αυτή τρομοκρατική δικαιολογία και στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν σε κρίσιμο σημείο οι σχέσει με, με τον ΝΑΤΟ, κοιτώντα και τα μηνύματα από την από Ανατολή, από τη Βόρεια Κορέα. Τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Να σα υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ήταν ε, ένθερμο υποστηρικτής των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ και είμαι, είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία. Να ακούσουμε και τις δικές σας ασφαλώ απόψει, κύριε Γενική Γραμματέα, για τι πρόσφατε εξελίξεις σε διεθνέ ε, προσκήνιο και το πώ θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν το λόγο στο Γενικό Γραμματέο και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να κάνουμε μια συζήτηση. Και πάλι την τεράστια τιμή που βρίσκεστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Ευχαριστώ, Άννα, για αυτή σας ε, την ε, φιλοξενία που μου παρέχετε και που με καλέσατε. Την περασμένη φορά που ήρθα να απευθυνθώ σε εσά ήταν πριν τη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία, πέρσι τον Ιούλιο. Και τώρα επανέρχομαι τρεις εβδομάδες πριν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, θα ξανασυναντηθούν στις Βρυξέλλες αυτή τη φορά στις 25 Μαΐου. Και χαίρομαι μπορώ να σας πω ότι από όταν σας συνάντησα την προηγούμενη φορά, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν υπέγραψα την κοινή δήλωση μαζί με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρόεδρο Τάσκ στη Βαρσοβία τον Ιούλιο. Αργότερα με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη συμφωνήσαμε το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους σε 42 συγκεκριμένα μέτρα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενισχύουμε την συνεργασία αυτή βασισμένη στο γεγονός ότι δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και αντιστρόφως. Συνεπώς, ε, η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία λήψης αποφάσεων και προς τις δύο πλευρές. Σεβόμαστε τις ε, διαφορές ανάμεσα στις, ε, στις δύο αυτές οργανώσεις και ταυτόχρονα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι και οι δύο έχουμε πολλά να κερδίσουμε από μια πιο στενή συνεργασία. Παρόλο ότι τα μέλη μας δεν ταυτίζονται, γνωρίζουμε ότι πάνω από το 90% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης, μοιραζόμαστε την ίδια ε, έλλειψη σταθερότητας, την ίδια στάθεια προς τον Νότο, το ίδιο περιβάλλον ασφάλειας, ε, τα ίδια προβλήματα στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τις ε, ίδιες προκλήσεις από μια όλο και πιο παρούσα Ρωσία. Συνεπώς όλοι αυτοί είναι λόγοι για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Και αυτό ακριβώς έχουμε κάνει με την κοινή δήλωση και με, τις 42, και με τα 42 μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόζουμε. Αυτά τα 42 μέτρα ε, έχουν σχέση με την ε, κυβερνοασφάλεια, με την απάντηση σε υβριδικές απειλές, με επιχειρήσεις, με γυμνάσια και ασκήσεις κλπ. Και πράγματι σημειώνουμε πρόοδο. Η ύπατη εκπρόσωπος κυρία Μογκερίνη θα ενημερώσει το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Εγώ αντιστοίχως το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ πάλι τον Ιούνιο για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει και μετά το καλοκαίρι θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να οικοδομήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Το θετικό είναι ότι δεν εφαρμόζουμε μόνο συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε αλλάξει όλη την κουλτούρα και την οτροπία της συνεργασίας μας. Η συνεργασία είναι πλέον ο κανόνας στις σχέσεις ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα ήταν η εξαίρεση πιο πολύ. Οπότε, να σας πω ότι ήδη έχει ενισχυθεί η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ανέβει ποιοτικά και ποσοτικά. Και ε, αυτό είναι το μήνυμά μου στους Υπουργούς Αμήνης. Ήταν το μήνυμά μου στους Υπουργούς Αμήνης την περασμένη εβδομάδα στη Μάλτα. Τους είπα ότι έχουμε ορατά και σαφή παραδείγματα συνεργασίας στη Μεσόγειο. Έξω από τις ακτές της Μάλτας, ήδη. Η, η επιχείρηση ασφάλειας στη θάλασσα Sea Guardian παρέχει προστα... Ε, υποστήριξη στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σοφία την περασμένη εβδομάδα τέσσερα πλοία του ΝΑΤΟ, τρία ε, αεροσκάφη ε, επιτήρησης θάλασσας βοήθησαν ε, την επιχείρηση Σοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συνεργαζόμαστε στο Αιγαίο με παρουσία σκαφών του ΝΑΤΟ προκειμένου να βοηθήσουμε να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, για να μειωθούν οι ροές παρανόμης μετανάστευσης. Αυτά δεν είναι μονολόγια, είναι πράξεις. Παραδείγματα πραγματικής και απτής βελτίωσης συνεργασίας. Κάτι που θα συνεχιστεί. Όπως σας είπα, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στις 25 Μαΐου εδώ στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση αυτή θα είναι σύντομη αλλά εξαιρετικά σημαντική. Για πρώτη φορά θα παραστεί ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα έρθει στην Ευρώπη, θα έρθει στο αρχείο του ΝΑΤΟ και για πρώτη φορά θα έρθει επίσης ο νέος Γάλλος πρόεδρος. 25 Μαΐου λοιπόν αυτή η συνάντηση θα είναι μια συνάντηση που θα στείλει ένα ισχυρό ηχηρό μήνυμα ενότητας, διατλαντικής ενότητας. Και μόνο η διοργάνωση και ε, το γεγονό ότι θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση μεταξύ των 28 και μάλιστα όχι 28, 29 γιατί θα έχουμε και το Μαυροβούνιο παρόν. Θα γίνει το 29ο μέλος της συμμαχίας. Ε, μόλις τα, όλα τα κοινοβούλια σε μερικές εβδομάδες θα έχουν επικυρώσει την ένταξή του. Τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν στην σύνοδο αυτή κορυφή του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ επίκαιρα και έχουν άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είτε είναι μέλη του ΝΑΤΟ είτε όχι. Πρώτον, ε, η κατανομή βαρών στην Διατλαντική Συμφωνία και δεύτερον, ο αγώνα κατά τη τρομοκρατία. Να τα σχολιάσω εν συντομία, χωρίς να επεκταθώ σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της ατζέντα του ΝΑΤΟ. Αν θέλετε θα μου υποβάλλετε ερωτήσεις για τα υπόλοιπα. Συνεπώς θα καλύψω τα πιο βασικά ζητήματα. Αυτά τα δύο ακριβώ ζητήματα που μόλις σας ανέφερα. Πρώτον, η καταπολέμηση τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία είναι μια υπαρκτή απειλή. Ε, ήδη λαμβάνουν χώρα και στι Πολιτείε, αλλά και στι πρωτεύουσε ε, των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιθέσει, τρομοκρατικέ επιθέσει ε, και αποτελούν πραγματικά επιθέσει εναντίον ανοιχτών δημοκρατικών κοινωνιών. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν μια ε, βεντάλια, ένα εύρος μέτρων, διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά, μέτρα που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια. Ε, κάποια από αυτά ε, είναι ε, μη στρατιωτικά, δεν έχουν καμία σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά κάποια άλλα, κάποια άλλα μέτρα ε, είναι στρατιωτικά και θα είναι στρατιωτικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την στρατιωτική πτυχή της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Στο Αφγανιστάν το είδαμε και το βλέπουμε και στην, στον αγώνα κατά του ISIS στο Ιράκ και τη Σύρια. χρειάζεται μια στρατιωτική πτυχή το ΝΑΤΟ έχει παίξει και συνεχίζει να παίζει ένα ρόλο κλειδί σε αυτά τα μέρη του κόσμου χρησιμοποιώντα στρατιωτικά μέσα. Στο Αφγανιστάν παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο για πολλά χρόνια. Η σημερινή μα, ε, ή μάλλον η στρατιωτική μα παρουσία στο Αφγανιστάν ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση του ΝΑΤΟ ποτέ. Συμμετείχαν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ και πολλά μη μέλη, πολλέ χώρε που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. στην επιχείρηση ISAF, για παράδειγμα, στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν είχαμε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση που δεν ήταν μέλη του ΝΑΤΟ. Κοινή λοιπόν αυτή η προσπάθεια και πρέπει να συνεχίσουμε την παρουσία μας εκεί. Δεν ε, ε, ε, έχουμε πολεμική δραστηριότητα πλέον εκεί, αλλά βοηθούμε, συνδράμουμε τις ε, ένοπλες δυνάμεις του Αφγανιστάν να ε, λάβουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και ένα από τα μαθήματα που μάθαμε από τα διδάγματα του Αφγανιστάν, αλλά και της, από τη Βοσνία Ζεγοβίνη και από το Κωσυφοπέδιο, είναι ότι μακροπρόθεσμα είναι πολύ καλύτερα ε, να ε, γυμνάζουμε τις τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις να χειρίζονται μόνες τους τη κατάσταση αντί εμείς να κάνουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, ανεξάρτητα. Επίσης πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για το τι είδους παρουσία θα έχουμε στο Αφγανιστάν τα επόμενα χρόνια. Καθώς επίσης και για το πώς θα ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξής μας στην ε, συμμαχία που έχουν ε, ιδρύσει οι Ηνωμένε Πολιτείε κατά του ISIS στη Συρία και το Ιράκ. Ε, εμείς ε, γυμνάζουμε αξιωματικούς του Ιράκ ως τώρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Χωρίς να εμπλακούμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μέσω μιας διαδικασίας που θα είναι πιο απαιτητική, θα πάρει πιο πολύ χρόνο ε, και που είναι η βοήθεια που θα πρέπει να δώσουμε στο Ιράκ και τις άλλες χώρες περιοχής να σταθούν από μόνες τους στα πόδια τους. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με πολλές από τις χώρες της ε, περιφέρειας αυτής για να τις σταθεροποιήσουμε. Το άλλο βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί στις 25 Μαΐου είναι και αυτό ένα θέμα στο οποίο έχουμε περιθώρια περισσότερη συνεργασία. Ε, εσείς έχετε πολλά εργαλεία, πολλά μέσα, έχουμε και εμείς δικά μας μέσα, ε, δεν τα έχει όλα, οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεργαστούμε και να τα θέσουμε σε κοινή χρήση. Το άλλο σημαντικό θέμα λοιπόν που θα συζητηθεί στη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων το Μάιο είναι ο διαταλικός σύνδεσμος και ο επιμερισμός προσπαθειών. Το ΝΑΤΟ στην Ουαλία το Σεπτέμβριο του 2014 πήρε μια απόφαση να σταματήσουμε τις μειώσεις στις στρατιωτικές μας δαπάνες, να τις αυξήσουμε σταδιακά και να φτάσουμε ε, σταδιακά στο 2% του ΑΕΠ στρατιωτικές δαπάνες στο τέλος της δεκαετίας. Το, η καλή είδηση είναι ότι ε, έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Μετά από πολλά έτη μειώσεων στις στρατιωτικές δαπάνες, το 2015 ήδη είδαμε μια μικρή αύξηση. Αμέσως μόλις αποφασίστηκε να σταματήσουν οι μειώσει και να περάσουμε σε αυξήσει. είδαμε ήδη από το 2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά μια αύξηση. Το 2016, τη δεύτερη χρονιά μετά την απόφαση, είδαμε μια σημαντική αύξηση στις στρατιωτικέ δαπάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. 3,8% του ΑΕΠ σε πραγματικού όρου. Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή. Σημαντική αύξηση. Οπότε κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάλι έχουμε πολλά περιθώρια βέβαια. Ε, γιατί ε, κάποιοι συμμαχοί είναι πολύ κοντά στο 2%, άλλοι το έχουν φτάσει, ενώ άλλοι είναι αρκετά μακριά από το 2%. Παρ' όλα αυτά κινούμαστε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατανομή των βαρών δεν έχει όμως σχέση μόνο με τις ε, δαπάνες. Έχει σχέση και με τις ικανότητες, τους πόρους. Χρειαζόμαστε πιο σύγχρονα όπλα, πιο σύγχρονες ικανότητες για, ε, να, ε, για να είμαστε πιο ισχυροί αποτρεπτικά. Το σημαντικό δεν είναι να επιλύουμε εκ των υστέρων της κρίσης, αλλά να τις αποτρέπουμε. Χρειαζόμαστε επίσης ε, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που έχουμε ήδη στήσει, πολλές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων το Μάιο. Ένα τμήμα της κατανομής των βαρών έχει σχέση με τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ξαναυπογραμμίσω ότι η ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα είναι κάτι το οποίο επιθυμεί το ΝΑΤΟ. Είναι καλή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλή για την Ευρώπη και είναι καλή και για το ΝΑΤΟ. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει πως αυτά που πράττει είναι συμπληρωματικά εναντί της δράσης του ΝΑΤΟ και δεν την ανταγωνίζονται. Αυτό είναι μια δέσμευση την οποία έχουν αναλάβει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας ε, συνεπάγεται μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες, περισσότερα γυμνάσια και ασκήσεις, περισσότερο εξοπλισμό και περισσότερη συνεργασία. Αλλά όχι προκειμένου να δημιουργηθούν καινούρια στρατηγία, ευρωπαϊκά στρατηγία τα οποία θα είναι, κινούνται παράλληλα με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ κλπ. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη δείχνουν ότι δεν θέλουν να ανταγωνίζονται, θέλουν να συνεργαστούν και το χρειαζόμαστε αυτό για να δημιουργηθεί μια άμυλα και όχι ένας ανταγωνισμός. Περισσότερο από το 90% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Το επαναλαμβάνω. Συνεπώς δεν έχει νόημα να ανταγωνιζόμαστε του εαυτούς μα. Οπότε το μήνυμά μου προς εσάς είναι ότι το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται σε, ένα περιβάλλον ασφαλείας πιο απαιτητικό. Ήδη ε, έχουμε, κάνουμε τις περισσότερες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και τη ε, μεγαλύτερη προσαρμογή όλων των τελευταίων δεκαετιών, αλλά χρειαζόμαστε με καλύτερη συνασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσουμε καλύτερα στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, τις οποίες ε, μοιραζόμαστε είτε είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στόλτενμπερκ για την παρουσίασή του. Και πρώτα απ' όλα τώρα θέλω να δώσω το λόγο στην πρόεδρο της Υποεπιτροπής, την κυρία Φωτίγκα, και στη συνέχεια στην κυρία Φακάλη, στην κυρία Κάλη. Καλή. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Αγαπητέ γραμματέα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την συνεχή θέλησή σας να ανταλλάζετε πληροφορίες και πρακτικές. Πραγματικά εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία σας και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των μελών της ε, Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Θα ήθελα να ξεκινήσω προσφέροντας τα συλληπιτήριά μας αλλά και την ανησυχία μας εξαιτία των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα σήμερα στην Καμπούλ και στόχευαν τα αρχηγεία της αποστολής στην Καμπούλ. Οκτώ Αυγανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους, καθώς και πάμπολοι στρατιωτικοί, αλλά και πολίτες μέλη της αποστολής συμπεριλαμβανομένων και τριών Αμερικανών στρατιωτών. Θέλω λοιπόν να σας εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου και στις οικογένειες του. Συχνά αναφέρουμε τα ζητήματα ασφαλείας εδώ στην Ευρώπη, αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν, οι περιοχές αυτές ζουν μέσα στη βία και συνεπώς η συμβολή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ καθώς και οι αποστολές πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύσσονται εκεί έχουν τεράστια σημασία. Και θέλω να θέσω εγώ προσωπικά ένα ερώτημα και να σας ζητήσω να αναπτύξετε περιττέρω την παρούσα κατάσταση στο Αφγανιστάν και να αναφερθεί τελείως στις αναγκαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις θητείες των αποστολών εκεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην παρούσα κατάσταση. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω ακόμα ποια είναι τα σχέδιά σας σε ό,τι αφορούν την ανατολική πτέρια του ΝΑΤΟ. Ε, τέλος, πρόσφατα σε διάφορες συνεδριάσεις ε, επιτροπών που έλαβαν χώρα στην Μάλτα παρουσία εκπροσώπων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αποστολών υπό την ηγεσία του κ. Μακάλιστερ παρακολουθήσαμε τα σχόλια της Φεντερίκα Μογκερίνη σχετικά με την ανάγκη να εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας στην Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των ε, διακινητών ανθρώπων, αυτών που πραγματικά εποφελούνται από παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Θα μπορούσατε λίγο να μοιραστείτε τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα και λίγο να ίσως να μας πείτε πώς θα μπορούσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτήκα και κυρία Καϊλή τώρα. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Αντιπροσωπεία ε, στην ε, κοινοβουλευτική συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα και εγώ να σα καλωσορίσω εδώ στη συνεδρίασή μα και κρυμώ ιδιαίτερα τον ενδιαφέρον σα για την τακτική ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα σε τέτοιε εποχέ μεγάλη αναστάτωση στην Ήπειρό μα. Θεωρούμε ότι οι ευρωβουλευτέ ε, συμβάλλουν απαραίτητα στην ε, διατήρηση των αξιών μας, στην προάσπιση των ζητημάτων μας σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όπως υπογραμμίσατε σε πολλές περιστάσεις και στην παρέμβασή σας. Το, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, πιο πολλές από παντού, από ποτέ, ε, και στην ε, γειτονιά μας ε, και στην ε, νότια γειτονιά, τη Λιβύη, Συρία, Ιράκ, στα Δυτικά Βαλκάνια, στάθειες και τριβές και προσφάτως ακόμα περισσότερη αστάθεια και νέες μορφές υβριδικού, κυβερνητικού πολέμου, κυβερνοπολέμου. Έχουμε την ρητορική της Τουρκίας, η οποία επίσης είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Έχουμε και το Brexit το οποίο σημαίνει ότι θα μας λείψει ο εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα είναι στον άτομο τουλάχιστον. Έχουμε και την τρομοκρατία, την μετανάστευση, όλα αυτά δεν γνωρίζουν σύνορα. Αυτές οι περίπλοκες λοιπόν προκλήσεις ζητούν και απαιτούν ε, περιπλοκές απαντήσεις, σύνθετες απαντήσεις και χρειάζονται λοιπόν η τυρική σχέση και υπάρχει πραγματικά αυτή η ανάγκη συμπληρωματικότητας προκειμένου να αποφευθούν οι αλληλεπικαλύψεις όπου αυτό είναι περιττό και σε δράσεις και σε δομές προκειμένου οι δαπάνες να είναι πιο αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να ενημερώσω και τους συναδέλφου μας εδώ ότι προσβλέπουμε στην έκθεση του Ιουνίου για την εφαρμογή της διακήρυξης της Βαρσομπίας για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και το κοινό πακέτο προτάσεων θα προσπαθήσουμε και πιο ενεργά να συμμετέχουμε στην ε, ε, Γεωργία σε ό,τι αφορά την διάσκεψη ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε πιο καθιερωμένες και πιο σωστές δομημένες σχέσεις, καλύτερη συνεργασία και όπως είπατε η συνεργασία είναι ο κανόνας πλέον και όχι η εξαίρεση. Θα ήθελα στη συνέχεια να υπογραμμίσω τον ε, ρόλο των βουλευτών στο ΝΑΤΟ και στην παροχή ε, ασφάλεια στους πολίτες για να υπάρξουν και μεγαλύτερες δαπάνες όπως τονίσατε προκειμένου να είναι Σημαντικό ο αντίκτυπο σε σχέση με τι θέσει τι οποίε εκπροσωπούμε. Θα ήθελα να σας θέσω δύο-τρεις ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Μία ερώτηση, καταρχάς, η κυβερνό άμυνα μας απασχολεί όλους. Δεν γνωρίζει σύνορα, όπως δεν γνωρίζει σύνορα και τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ απαραίτητο να ανταλλάσσουμε ε, πληροφορίε. Ένα από του επτά στόχου. Ε, που έχουμε θέσει για τη συνεργασία, για ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών για την κυβερνοάμυνα. Ρωτώ λοιπόν, ενημερώστε μα, τι πρόοδος ε, έχει σημειωθεί στον στόχο αυτό από πλευρά του ΝΑΤΟ και ε, τι πρόοδος υπάρχει για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σύμμαχων. Ε, αναμένεται καμία έκπληξη επίση στι 25 Μαΐου Αυτές ήταν οι βασικές ερωτήσεις επί του παρόντος ε, και μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια και στη Γεωργία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την κυρία Φωτίγκα, ευχαριστούμε και την ε, κυρία Κάιλη. Έχουμε ε, μία ώρα ακριβώς μέχρι τις 4.30 και 25 άτομα που έχουν ζητήσει τον λόγο. Καταρχάς, δύο λεπτά maximum ο καθένας Πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Άτεκτος. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Όχι δύο και δεκαπέντε, όχι και δύο και δέκα. Και σε δεύτερη φάση θα ακούσουμε όσο πιο πολλού συναδέλφου γίνεται και μόλι ο κύριο Τότλεμπερ μα πει «Δεν μπορώ άλλο» φτάνει, τότε θα σταματήσουμε για να ακούσουμε τι απαντήσει. Και παρεμπιπτόντω δεν χρειάζεται να εξαντλήσετε τα δύο λεπτά αυτά, είναι το όριο να ξεκινήσουμε με τον Μίχελ Γκάλ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώ ορίσατε και στην Επιτροπή μα. Ένα από του λόγου για του οποίου και εγώ συγκαταλέγομαι μεταξύ των όσων ε, προασπίζονται συμπληρωματικέ, αλλά και αυτόνομες στρατιωτικές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ένα από τα πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, η Τουρκία αναφέρθηκε, που δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δικαίωμα αρνησυγκρίας, βέτο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όπως όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ άλλωστε. Και γι' αυτό πιστεύω για να γλιτώσουμε από αυτό ενδεχομένως θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε δυνατότητα να δρούμε ανεξάρτητα σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη γεωγραφικός πώς, ε, όπου θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να δράσουμε, ενώ η Τουρκία μπορεί να μην το θεωρεί αυτό απαραίτητο και να προβάλλει βέτο. Έχετε οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη ότι η Τουρκία εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται. Ατυχώς πως αυτό επηρεάζει την ε, συμπεριφορά της όμως στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Αυτό αφενός, αφετέρου. Ξέρουμε ότι πολλοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο γιατί δεν ξέρουν ποια θα είναι η μοίρα του όταν θα επιστρέψουν στην χώρα του. Εσεί, ασφαλώ, ω ΝΑΤΟ δεν μπορείτε να χορηγήσετε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει κάποια δραστηριότητα από κρατημέλη τα οποία ενδεχομένω να είναι τεθειμένα να του δεχτούν. για να μην βρεθεί κανεί από τον ΝΑΤΟ κατευθείαν στη φυλακή όταν επιστρέψει στη χώρα του. Τελευταία ερώτηση. σε κάποιες περιπτώσει υπάρχουν ισχυρισμοί ότι υπάρχουν παράλληλες δομές. κοιτώντα τι αποστολές που έχουμε στο κέρα της Αφρικής ω Ευρωπαϊκή Ένωση, ω ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο, η Σοφία και αυτά που κάνει το ΝΑΤΟ, δεν θα είχε νόημα μήπω πριν από την επιχείρηση αυτή να συμφωνούμε ότι θα το κάνει αυτό η μία ομάδα ή η άλλη ομάδα. Διαζευτικά. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα είχε πιο μεγάλο αποτέλεσμα, θα ήταν πιο αποδοτικό. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ακριβώ. Ο Κνούτ Φλέκενστάιν από του Σοσιαλιστέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα. Δεν έχω καμία ερώτηση να κάνω. Εγώ μόνο δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω από δική μα πλευρά. Το πρώτο. Η κατανομή των καθηκόντων. Το θέμα δεν είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί με τους δε. Το θέμα είναι να πετύχουμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα ε, ως καλή εταίροι μέσα στο ΝΑΤΟ ή του ΝΑΤΟ. Καταρχάς, δεδομένου και των νέων προκλήσεων που ανακύπτουν, να αναλαμβάνουμε καθήκοντα τα οποία θα προστίθονται επιπροσθέτως προς τα παλιά καθήκοντα και κατά δεύτερον να συμβάλλουμε προκειμένου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ενδεχομένως να μπορούν να μπορούν ε, με την κοινή του ε, εργασία να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να επιτελούν τα καθήκοντα τους πιο αποτελεσματικά έως τώρα. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ είναι το εξή. Ε, το θέμα του burden sharing, του επιμερισμού των καθηκόντων. Νομίζω ότι όλοι εδώ ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολλά από αυτά που έχουμε κάνει έως τώρα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και επίσης είναι σημαντικό, θεωρώ, να επικεντρωνόμαστε πάντα σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, επιπροσθέτως. Και οι πιο πολλές δαπάνες για το στρατιωτικό σκέλος θεωρώ ότι δεν αποτελεί κάποιο κατόρθωμα, κάποιο επίτευγμα. Το θέμα είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τα μέσα που ήδη διαθέτουμε. Τι να τα κάνουμε τα γερμανικά αεροσκάφη άμα δεν πετάνε. Μην σας πω ότι κοστίζουν και πάρα πολλά χρήματα. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι χρειάζεται αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και σε μεγαλύτερο βαθμό θα χρειαστούν και παραπάνω δαπάνες, ναι. Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατανομή των ευθυνών, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε και το εξή. Συμπεριλαμβάνει αυτό και τη δουλειά που α, κάνουμε στον πολιτικό σκέλος, αναπτυξιακή βοήθεια και το καθεξής. Άρα το 2% θεωρώ ότι δεν είναι το μέτρο που μετράει. Η κατανομή των πραγματικών καθήκοντων είναι το σημαντικό. Ο κύριος Τάνοκ από το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, με χαρά μου ακούω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, ε, όπως η αλληλεπικάλυψη, και λοιπά δεν ε, ισχύουν πλέον και μπορούμε πλέον να συνεργαστούμε προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης απειλών όπως το ISIS, η Ρωσία κλπ. Χαίρομαι που το Μευροβούνιο ε, είναι ε, σχεδόν μέσα στο ΝΑΤΟ. χαίρομαι που θα έρθει ο κύριος Τραμπ εδώ. Βέβαια, η Ελλάδα, η Εστονία και η χώρα μου έχουν ξεπεράσει το 2%. Ε, με χαροποιεί αυτό. Αυτό με χαροποιεί είναι ότι ο κ. Τραμπ θα συναντήσει τον ε, πρόεδρο τη Βόρεια Κορέα. Ε, η, το Ηνωμένο Βασιλείο θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα υιοθετήσουμε το νορβηγικό μοντέλο σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ και ότι θα μείνουμε ε, κοντά στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και την κοινή, εξωτερική, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι επίσης θα ε, υιοθετήσουμε το ε, στρατιωτικό δόγμα της Σουηδίας που ε, έχει ε, υπογράψει, έχει δεσμευθεί μάλλον στην τήρηση του άρθρου 5 περί προάσπισης των συνόρων των γειτόνων της, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ελπίζω επίσης ότι το 42-7 και το 2.22 της, ε, της ε, Συμφωνίας της Λισαβόνας θα τηρηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά την έξοδό της ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να, ξα... να μείνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ καλοί σύμμαχοι. And now we come to Mrs. Κυρία Βάλτμαν, από τους φιλελεύθερου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα μιλήσω Ολλανδικά. Ναι, ναι, ναι, να βάλετε τα ακουστικά σα θα περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και χαίρομαι ιδιαίτερως που στην αρχή τη παρέμβασής σα είπατε ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ είναι πλέον ο κανόνα ενώ παλαιότερα ήταν η εξαίρεση. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο και νομίζω ότι από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούμε παρά να το χειροκροτήσουμε. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να κοιτάξουμε μαζί. Καταρχά, όταν ε, ο νέο πρόεδρο τη Αμερική ε, εκλέχθηκε πριν από κάποιο καιρό, ε, είχαμε μείνει λίγο άναυδοι. Σοκαριστήκαμε από τις δηλώσεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης ε, δεν θα μπορούσαμε πλέον να υπολογίζουμε στο ΝΑΤΟ, γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Ε. Αλλά αυτό που πρέπει να παρατηρήσω είναι ότι αυτό δεν υλοποιήθηκε ευτυχώς. Εσείς πώς τοποθετήσετε εναντί των δηλώσεων του Προέδρου του ΙΠΑ και πώ θα τοποθετηθείτε στην επόμενη συνέβα του ΝΑΤΟ. Δεύτερο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό για μα, το αναφέρατε κι εσεί άλλωστε ήδη, τι θα κάνουμε με τη Ρωσία. Η Ρωσία παραμένει μια χώρα γειτονική τη Ευρώπη. Πολύ δύσκολε προ το παρόν οι σχέσει. Πολύ δύσκολε οι σχέσει με τη Ρωσία και αναρωτιέμαι τι είδου στρατηγική θα ακολουθήσει το ΝΑΤΟ στο μέλλον έναντι της Ρωσίας. Τρίτο, και το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, η Τουρκία. Χθε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έγκριναμε κι άλλη μια έκθεση πρόοδου, πρόοδου, ο Θεός να την κάνει πρόοδο μάλλον, οπισθοχώρησης και καταλήγουμε στο ότι δεν μπορεί να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα την αντιμετωπίσουμε όμω στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και αυτό είναι σημαντικό. Τέλος, οι Ευρωπαίοι πολίτε ζητούν στι τελευταίε δημοσκοπήσεις του Μέτρο να βάλουμε κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια. Το είπατε ότι και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατία. Ερωτώ λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα κατά της δημοκρατίας μαζί με το ΝΑΤΟ και με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Και τώρα να περάσουμε στην κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το αρχηγείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης του ΝΑΤΟ. Το αρχηγείο για την εφαρμογή μη εκτελεστικών αποφάσεων. Παλιά πολλά κράτη του ΝΑΤΟ και κυρίως η ΙΠΑ ήταν κατά ενός τέτοιου αρχηγείου. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πλέον δεν ισχύει. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι η υποστήριξη αυτή θα συνεχιστεί σε περίπτωση που θα υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια για την επέκτηση των αρμοδιοτήτων του αρχηγείου και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άλλη μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την κοινή, τα κοινά συγκεκριμένα σχέδια και έργα. 42 συγκεκριμένα σχέδια προγραμματίζονται. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Να συνεχίσω. 42 λοιπόν κοινά τέτοια έργα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ προγραμματίζονται. Πολλά εξ αυτών από ό,τι είπατε θα λάβουν χώρα και στη Μεσόγειο και αναφέρατε ε, ως παράδειγμα την επιχείρηση Σοφία. Ρωτώ, υπάρχουν άλλα σχέδια για άλλες περιοχές στις οποίες θα λάβουν χώρα θαλάσσιες επιχειρήσεις. Άλλη ερώτηση. Η επέκταση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε τι βαθμό περιλαμβάνει και ουδέτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιρλανδία. Συζητιέται το θέμα αυτό, κατά πόσον δηλαδή αυτό συμβαδίζει με την ουδετερότητα των κρατών αυτών, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει μεγαλύτερη συμμαχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Βαλέρο, από τους Πράσινους. Eh, Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την ε, συνεργασία στην Μεσόγειο. Γιατί δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τη μετανάστευση με στρατιωτικά μέσα, δεν είναι ποτέ δυνατόν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι για την μετανάστευση, ενώ πρέπει να σώσουμε κόσμο στην Μεσόγειο. Αυτό είναι που κάνουμε. Και ίσως αυτό να μην είναι ο πρωταρχικός στόχος του ΝΑΤΟ σε κάθε περίπτωση. Και θέλω να ρωτήσω κάτι και για τον στόχο του 2%. Βεβαίως η Σουηδία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επομένως δεν έχουμε τη δέσμευση αυτή. Όλες οι άλλες χώρες όμως την έχουν. Η ερώτηση είναι τι αγοράζουμε με αυτό το 2%. Πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να έχουμε με αυτό το 2%, όχι τι ποσοστό θα πρέπει να συνεισφέρουμε. Αλλά όπως είπε και ένας συνάδελφος, υπάρχουν πολλά σχέδια αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αν δεν έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό. Το να αγοράσουμε εξοπλισμό χωρίς να έχουμε την ποιότητα που πρέπει να έχει ο, το, ο αμυντικός μας εξοπλισμός, τι μας προσφέρει. Και υπάρχουν αρκετά διαφορετικά σχέδια που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε χρήματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ό,τι αφορά τα αμυντικά συστήματα των διαφόρων κρατών μελών αντί να αυξάνουμε τις ε, δαπάνες συνεχώς. Επομένως, δεν είναι απλά ζήτημα ποσοτικό αυτό το 2%. Είναι ανάγκη να κοιτάξουμε λίγο την ποιότητα. Είναι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει στην άμυνα, όχι απαραίτητα η ποσότητα. Ευχαριστούμε. Κανένας από το EFTD δεν θέλει να μιλήσει. EFTD. Όχι, κύριε Σάφερς, εσείς δεν είστε EFTD, εκτός και αν έχετε αλλάξει κόμμα και δεν μας έχετε ενημερώσει. Περνάμε τώρα στο ENF και ο κύριος Μποργέζιο είναι ο πρώτος ομιλητής. Με έχουν ε, ενημερώσει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με τον Ιταλικό με την Ιταλική καμπίνα. Μπορείτε να μιλήσετε Ιταλικά και θα, έχετε, θα υπάρχει διερμηνία, αλλά δεν υπάρχει κανείς να... δεν μπορείτε να ακούσετε Ιταλικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπογραμμίσατε ότι υπάρχει μια πρωταρχική δέσμευση του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την ανάγκη αναχέτηση των μεταναστευτικών ε, ροών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα η, η μάχη αυτή να, να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω το εξής. Γνωρίζετε πολύ καλά την Μεσόγειο, έχετε γίνει ειδικό των διαδρομών, αυτών των θαλάσσιων διαδρομών, ιδιαίτερα σημαντική για τους διακινητές, για τους παράνομους διακινητές μεταναστών. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια τρομερή μια περίπτωση που αφορούσε τις Ιταλικές αρχές με αρκετά σκιώδεις περιπτώσεις χρηματισμών και συνομιλίες με διακινητή. Υπήρχαν ύποπτοι στην υπόθεση αυτή. Υπήρχαν επίσης διασυνδέσεις διείσδυσης τρομοκρατών. Γνωρίζετε ίσως ότι η πλειοψηφία των πλοίων από την Λιβύη ελέγχονται από τους τζιχαντιστές. Και πώς το ΝΑΤΟ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα αυτή, την οποία κατήγγυλαν, επαναλαμβάνω, κατήγγειλε ο Ισαγγελέα στην Ιταλία, μια ανεξάρτητη περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μποργέζιο που μίλησε στα γαλλικά. Έχουμε έναν ακόμη ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, μας αναφέρατε προηγουμένως ότι το ΝΑΤΟ θέλει μια στρατηγικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή τη στιγμή από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο δύο, η Ελλάδα και η Κύπρος, υφίστανται πραγματική απειλή αυτή που προέρχεται από την Τουρκία. Γνωρίζετε πολύ καλά εχθές ότι εχθές συγγνώμη, ο πρόεδρος Ερδογάν απείλησε πρώτα την Κύπρο και μετά την Ελλάδα ότι αν επιτρέψουν σε διεθνείς εταιρείε να κάνουν έρευνες για εξόριξη πετρελαίου και αερίου στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χώρων αυτών θα τους κηρύξει πόλεμο. Τους απείλησε δηλαδή με κάζους μπέλη και έστειλε και σχετικό έγγραφο στον ΟΗΕ. Συνεπώς για τις δύο αυτές χώρες είναι λογικό, αναμενόμενο και επιβεβλημένο να έχουν υψηλές στρατιωτικές δαπάνες. Για τις υπόλοιπε όμως χώρες, για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η υποχρέωση. Ποιος είναι ο πανίσχυρος εχθρός, ο οποίος απειλεί τον ΝΑΤΟ και ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο τεχνοκρατικά, αυτή τη στιγμή τα στρατιωτικά επιτελεία του ΝΑΤΟ ποια σχέδια επιχειρήσεων συντάσσουν εναντίον τίνος εχθρού, καθώς επίσης και ποια σχέδια ενδεχομένων επιχειρήσεων, τα contingency plans όπως θα ξέρετε, ε, σχεδιάζονται εναντίον ποιου εχθρού, με ποιες δυνάμεις και κατά πόσον πρέπει να ενισχυθούν πραγματικά οι δυνάμεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα, αυτό ήταν ο πρώτο γύρο λοιπόν ερωτήσεων και τώρα, Γενική Γραμματέα, από σα εξαρτάται ε, να χρησιμοποιήσετε όσο χρόνο θέλετε για να απαντήσετε. Σα υπενθυμίζουμε απλά γενικά ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να θέσουν ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για τι ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα πιο βασικά ζητήματα τα οποία θίξατε. Ενδεχομένω να μην μπορέσω να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει, γιατί προφανώ κάποιε. Ε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για την ε, τα συλληπιτήρια που εκφράσατε για όσους χάσαν τη ζωή τους ή την οικογένειά τους στη σημερινή επίθεση στην Καμπούλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στον Αφγανιστάν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να συνεχίσει να είναι εκεί το ΝΑΤΟ. Όχι στις ενόπλες, ε, στον ενόπλο αγώνα, αλλά για την εκπαίδευση και την παροχή βοήθεια στους Αφγανούς για να αντιμετωπίσουν τις τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις, όπως η σημερινή. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει ακόμα για να αλλάξει η εντολή τη αποστολή. Το θέμα δηλαδή είναι η εκπαίδευση και η παροχή αρρωγή, όχι η στρατιωτική ανάμειξη. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία. Και αργότερα, μέσα στο χρόνο, θα το συζητήσουμε αυτό και το Μάιο και τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, μάλλον ζωτήσατε να σας πω για την καταπολέμηση της ε, μετανάστευσης. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από διάφορους ε, βουλευτές. Η μετανάστευση προαπαιτεί μία ανταπόκριση εθνών και μάλιστα εθνών και πολλών ε, παγκοσμίων οργανισμών. Ο ΙΕ, τα μεμονωμένα έθνη. Χρειάζεται μία απάντηση από όλα τα κράτη και από άλλους τους οργανισμούς. Εγώ τι μπορώ να κάνω, να πω το πώς μπορεί να συμβάλλει το ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας για να ανταποκριθεί στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Να θυμόμαστε βέβαια ότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία. Χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους και αυτό δείχνει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες διαβίωσης σε πολλές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ΝΑΤΟ βοηθάει εν μέρη καταπολεμώντας τις βαθύτερες αιτίε. Γι' αυτό προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε το Αφγανιστάν, προσπαθούμε να καταπολύσουμε την τρομοκρατία στο Ιράκ, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας όπως η Τινησία, η Ορδανία. Ο στόχος μας είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε όλη την περιοχή, μειώνοντας και τις αιτίες που προκαλούν την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια, τότε θα είναι όλο και πιο λίγοι αυτοί που φεύγουν από τις χώρες τους, γιατί θα είναι πιο λίγοι αυτοί οι οποίοι απειλούνται από τον πόλεμο και από τη βία, αλλά γιατί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη είναι προαπαιτούμενα για οικονομική ανάπτυξη ακόμα και αυτοί που δεν φεύγουν τη χώρα τους λόγω πολέμου, αλλά λόγω φτώχειας αν αντιμετωπίσουμε αυτές τις βαθύτερες αιτίε με δημιουργώντας ασφάλεια και ειρήνη, δημιουργούμε τη βάση για οικονομική ευημερία. Και αυτό διώχνει πολύ κόσμο. Δεν λέω ότι το ΝΑΤΟ είναι η απάντηση. Αυτό που λέω είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι τμήμα της απάντησης και έτσι συμβάλλουμε με διαφορετικούς τρόπους και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς προς αυτό το σκοπό. Η κυρία Καηλή. Να πω ότι καταρχά εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνατε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνέλευση για το ΝΑΤΟ και εγώ ήμουν βουλευτή για πάρα πολλά χρόνια, από το 1991. Ξέρω τη σημασία των κοινοβουλίων. Τα κοινοβούλια αποφασίζουν για την νομοθεσία, για το πλαίσιο τη πολιτική ασφαλεία και άμυνα και αποφασίζουν και για τη χρηματοδότηση, για τον προπολογισμό. Άρα, με καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ισχυρή πολιτική άμυνας και ασφάλειας χωρί την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη δουλειά που κάνετε. Οι βρυδικέ απειλέ. Συνεργαζόμαστε από αυτόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ασκήσεις που έχουν να κάνουν με τις υβρετικές απειλές και και απειλές και οτιδήποτε συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Με ρωτήσατε κατά πόσον αναμένω εκπλήξεις ε, στην συνάντηση στις 25 Μαΐου αρχήγων κυβερνήσεων και κρατών. Δεν αναμένω με εκπλήξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις εκπλήξεις άλλωστε. Δεν μπορεί να τις προβλέψει κανείς ποτέ. Εγώ δεν θέλω να υπάρξουν εκπλήξεις όμως. Ελπίζουμε να προγραμματίσουμε με τέτοιο τρόπο τη συνάντηση ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξει. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανεί τι θα προκύψει την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια, ο κύριο Γκάλερ. Συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία του ΝΑΤΟ και το πόσο τη σημασία να μπορεί να δρά αυτόνομα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ βεβαίω, βεβαίω. είμαστε, δύο ανεξάρτητοι οργανισμοί. Πώ να το κάνουμε. Έχουμε αυτόνομε διαδικασίε λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να λαμβάνουμε τι δικέ μα αποφάσει. Αλλά ασφαλώ και έχουμε μεγάλου συνδέσμου, γιατί έχουμε την ίδια γειτονία, έχουμε σε μεγάλο βαθμό τα ίδια μέλη. Και ακόμα και όσοι δεν είναι μέλη και των δύο οργανώσεων έχουν στενέ σχέσει. Έχουμε την Νορβηγία. Δεν είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σουηδία, η Φιλανδία δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά είναι εταίροι του ΝΑΤΟ όπως και η Αυστρία και η Μάλτα. Άρα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με πολλούς στενούς δεσμούς. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αυτονομία και τις διαφορές μεταξύ των οργανώσεων, αλλά να σεβαστούμε και τα κοινά μας στοιχεία να προσθέσω γιατί αυτό έχει να κάνει και με πολλές ερωτήσεις που μου θέσατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά εργαλεία τα οποία δεν έχει στην διάθεσή του το ΝΑΤΟ. Διπλωματία, οικονομικά εργαλεία, πάρα πολλά εργαλεία τα οποία εμεί δεν έχουμε στην διάθεσή μα. Εκ παραλλήλου, πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τη συλλογική άμυνα, ιδιαίτερα των συμμάχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει περίπτωση να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Και αυτό επίση εκφράστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Άμυνα δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την συλλογική άμυνα την οποία παρέχει το ΝΑΤΟ στου συμμάχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 80% των επενδύσεων των αμυντικών του ΝΑΤΟ θα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τρεις από τα τέσσερα τάγματα θα είναι υπογειοσία μη α, χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά, Καναδάς, Πολιτείε και Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες απόψεις για του συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά είναι σαφές ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την ασφάλεια της ε, ε, Ευρώπης. Η Αλβανία είναι τμήμα των προσπαθειών μας να σταθεροποιήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια σημαντικά για όλη την Ευρώπη και δείχνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Καναδά και της ΙΠΑ. Στο βορρά δε έχουμε και χώρες όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία. Άρα υπάρχουν ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το μήνυμα που έχω να στείλω είναι το εξή. Είμαστε αυτόνομε οργανώσει και πρέπει να είναι σεβαστέ σε διαφορέ, αλλά η συλλογική άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι κάτι το οποίο αποτελεί βασική ερμοδιότητα του ΝΑΤΟ. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι απάντησα σε διάφορε ερωτήσει ε, μόνο μια. Φλέκενστάιν. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και το θέμα της κατανομής των ευθυνών και της ε, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Το θέμα της αποτελεσματικότητας. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να δαπανούμε καλύτερα και πιο πολλά. Το θέμα δεν είναι να δαπανούμε πιο πολλά μόνο ή καλύτερα μόνο. Όχι. Και τα δύο συμφωνήσαμε το 2014 και αύξηση των εμπορικών των ε, στρατιωτικών δαπανών και καλύτερη αξιοποίηση των δαπανών αυτών. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολιτικοί θα ήθελαν να δαπανίσουμε στην ε, εκπαίδευση, την υγεία, στις υποδομές και όχι στην ε, άμυνα. Και όταν ήμουν υπουργό οικονομικών στη δεκαετία του 90 στην Νορβηγία, εγώ μείωσα τις τακτικές επενδύσεις, ε, τις επενδύσεις στην άμυνα. Ήταν μετά τον ψυχρό πόλεμο. Μετά τον ψυχρό πόλεμο και όλοι μείωναν τις επενδύσεις στην άμυνα. Και όταν τα πράγματα πάνε καλά, είναι λογικό να μειώνονται αυτές οι ταπάνες, θεωρώ. Αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε, να αυξάνουμε και τις ταπάνες αυτές όταν αυξάνονται και οι τριβές. Και τώρα λοιπόν ο Υπουργό Οικονομικών Θεωρών στην Νορβηγία είναι υπεύθυνο για να αυξήσει τι δαπάνε αυτέ. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση, μια και υπάρχουν μεγαλύτερε τριβέ. Τώρα, για το Brexit και το νορβηγικό μοντέλο. Καταρχά, δεν ξέρω τι να σα πω ακριβώ για το νορβηγικό μοντέλο. Για να είμαι και ειλικρινή, εγώ ήμουν ε, από του βασικού υπερμάχου τη συμμετοχή, τη ένταξη τη Νορβηγία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 που είχε γίνει ε, το δημοψήφισμα. Και είχα πει τότε ότι είχαμε διαπραγματευτεί σύμβαση ε, προσχώρησης δύο φορές, το 72 και το 94. Και μετά καταψηφίστηκε, όχι μία φορά, αλλά δύο, στο δημοψήφισμα η ένταξη στην ε, Ένωση. Άρα τι να σας πω, εγώ δεν είμαι υπέρ του νορβηγικού μοντέλου, ήμουν κατά του νορβηγικού μοντέλου, εγώ ήθελα να μπούμε στην Ένωση. Δεν τα κατάφερα, αλλά τι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ήθελα να έρθω και εδώ, γιατί ήταν το πιο κοντινό που μπορούσα να πετύχω σε ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι να κάνουμε, αφού δεν είμαστε μέλη Προφανώς ε, το νορβηγικό μοντέλο αυτό ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος θεωρώ ότι αποτελεί ένας καλός τρόπος για την ένταξη κάπως στην ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα. για τον Τραμπ και τις Αμερικανικές εκλογές. Καταρχάς, ήταν ε, συνεκτικό το μήνυμα του κυρίου του Πρόεδρου Τραμπ σε όλες τις συζητήσεις μου μαζί του ότι οι ΙΠΑ παραμένουν δεσμευμένοι στην Διατλαντική Συμμαχία και στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το μήνυμα όταν του μίλησα αμέσως μετά την εκλογή του. Αυτό ήταν και το μήνυμα όταν του μίλησα μετά την ορκομοσία του τον Ιανουάριο. Και αυτό ήταν και το μήνυμα όταν συναντήθηκα πριν από δύο εβδομάδες μαζί του στο Λευκό Οικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία 28 δημοκρατιών, όπου εκλεγμένοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων συζητάνε για πάρα πολλά διαφορετικά θέματα. Αλλά η, ισχύ, θέματα. Αλλά η ισχύ του ΝΑΤΟ είναι ότι επανελειμμένω μπορούμε να αποδείξουμε ότι παρά τι πολιτικέ αυτέ διαφορέ πάντα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε επί των βασικών στοιχείων του ΝΑΤΟ ότι είμαστε μαζί ενωμένοι, προστατεύουμε οι μεν του δε και αναγνωρίζουμε ότι είμαστε πιο ισχυροί ενωμένοι παρά ο καθένα ξεχωριστά. Ε, μία, ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για την Ευρώπη αλλά και για τι ΗΠΑ Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και ένας ψυχρός πόλεμος χρειάστηκαν για να κατανοήσουμε ότι αυτά είναι σημαντικά και για τον Καναδά και για τη ΣΥΠΑ και για τη Βορειοαμερική. Αμερική. Να θυμόμαστε επίσης ότι το μοναδικό, η μοναδική περίπτωση που έγινε επίκληση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ήταν μετά την επίθεση της ΙΠΑ. Ε, Στο Αφγανιστάν ε, χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους ε, στο Αφγανιστάν μετά από την επίθεση αυτή στην Αμερική. Αλλά ως, άρα ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το ΝΑΤΟ είναι σημαντικό για πολλούς Ευρωπαίους ε, συμμάχους, αλλά το ΝΑΤΟ είναι σημαντικό και για τη Βόρεια Αμερική. Ρωσία. Εν συντομία. Η Ρωσία. Ε, για θέματα άμυνας και διαλόγου. Αυξάνουμε την παρουσία μας ε, στην α, περιοχή αυτή όχι για να προκαλέσουμε τη Ρωσία, αλλά για να την αποτρέψουμε. Η εμπειρία μου ως πολιτικός είναι ότι δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ ισχύω και διαλόγου. Όσο είναι κανείς ισχυρός και είναι προβλέψιμος και έχει πολλούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ, μπορεί να μιλήσει στη Ρωσία. Αυτό κάνουμε και με στην Νορβηγία. Έχουμε ένα κοινό. Έχουμε κοινά σύνορα με τη Ρωσία, χερσαία και θαλάσσια. Αλλά έχουμε μια ρεαλιστική εύρυθμα λειτουργούσα συνεργασία και συζήτηση με τη Ρωσία. Όχι παρά το γεγονός ότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά επειδή είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα όσο είμαστε ισχυροί και δυνατοί, μπορούμε να κάνουμε πολιτικό διάλογο με τη Ρωσία. Η Ρωσία, ξέρετε, είναι γειτονά μας. Δεν πρόκειται να φύγει. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις εντάσεις και τις τριβές, να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν χαιρόμαστε που υπάρχει ο πολιτικό διάλογο, γιατί πρέπει να είναι πιο επικοδομητική η σχέση με τη Ρωσία. Για την Τουρκία, εν συντομία. Η Τουρκία είναι σημαντικό εταίρο. Μεταξύ άλλων και λόγω τη γεωγραφική τη θέση κοντά στο Ιράκ, τη Συρία, την ε, Ρωσία, στον Εύξηνο Πόντο. Κλειδί για την ε, μεταναστευτική αντιμετώπιση του, της μεταναστευτικής κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. διάφορες απόπειρες πέρσι τον Ιούλιο. Και φυσικά και η Τουρκία έχει δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό της κατά του πραξικο... της απόπειρας πραξικοπήματος. Αλλά να θυμόμαστε και τις βασικές μας θεμελιώδεις μας αξίες. Ε, δημοκρατία, κράτος δικαίου και το έχω συζητήσει αυτό σε διάφορες περιστάσεις, σε διάφορες πρωτεύουσε του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και στην Άγκυρα. Γιατί αυτές οι αξίες είναι σημαντικές για την συμμαχία και είναι σημαντικές και για μένα ως Γενικός Γραμματέος. Έχετε δίκιο ότι κάποιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, κάποιοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ζητήσει άσυλο. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουν τα μεμονωμενα κρατημέλη σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Κατά πόσον θα δεχτούν την αίτηση αυτή για άσυλο και κατά πόσον θα χορηγήσουν άσυλο. Δεν είναι ζήτημα του ΝΑΤΟ, δεν είναι καθήκον του ΝΑΤΟ να λάβει τέτοιε αποφάσει. Η κυρία Λούζινγκ Υπάρχει ένα σχεδιασμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μάλλον ένα αρχηγείο το οποίο θα δημιουργηθεί και θα ιδρυθεί. Δεν νομίζω ότι επαφείται σε μένα να σχολιάσω την εντολή του γραφείου αυτού. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χαιρετίζω το γεγονός ότι εκφράστηκε ξεκάθαρα ότι η αλληλεπικάλυψη αυτών των καθηκόντων είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Είναι διαφορετικό αυτό το γραφείο. Είναι διαφορετική αυτή η μονάδα σε σχέση με τα αρχηγεία του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα τώρα του κατά πόσο μπορούμε να σεβαστούμε τι ουδέτερε χώρε. Μα βέβαια, νομίζω ότι μία από τις, ε, ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ και η δύναμη του ΝΑΤΟ είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με ουδέτερε χώρε επί σειρά ετών. Η Σουηδία, η Φιλανδία, πολύ στενή εταίροι του ΝΑΤΟ και η Αυστρία άλλωστε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, ασκήσεις, σε δυνάμεις ε, στο Κωσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν. Είμαστε απόλυτα σε θέση να συνεργαστούμε με οδετρές χώρες. Ήμουν και στη Μάλτα προσφάτως, όπου και εξέφρασα ακριβώς το ίδιο. Οι εταίροι συχνά είναι ουδέτεροι και μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, σεβόμενοι απόλυτα την ουδετερότητά τους. για τη Σουηδία τώρα. Για τα θρησκευτικά μέσα και τη μετανάστευση. Τα θρησκευτικά μέσα ασφαλώς δεν αποτελούν την πρώτη αντίδραση στους μετανάστες. Αλλά τα στρατιωτικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την κρίση στο Αιγαίο, για παράδειγμα. Όπως αντιμετωπίζουμε με στρατιωτική ε, επιχείρηση στο Αιγαίο και προωθούμε τη συμφωνία την Τουρκία. Και έτσι αποτρέπουμε τον κόσμο από το να διασχίζει τη Μεσόγειο. Και έχουμε και την επιχείρηση Σοφία, για παράδειγμα. Το 2% τώρα. Θα συμφωνήσω και πάλι μαζί σα. ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο output, στο τι πετυχαίνουμε με το 2% αυτό. Και όχι μόνο στο πόσα χρήματα δαπανούμε, αλλά χρειαζόμαστε και παραπάνω δαπάνες, όπως σας είπα, και καλύτερη αξιοποίηση αυτών. Μποργέζιο. Είναι πολύ, πολύ σύνθετο το θέμα του προσφυγικού και των μεταναστών. Και πάλι χρειάζονται πάρα πολύ, πολλά εργαλεία τα οποία δεν είναι στρατιωτικά στη φύση του και πολλά τέτοια μέτρα εκτός του ΝΑΤΟ. Αλλά το ΝΑΤΟ βοηθάει με την παρουσία μα στο Αιγαίο, στην Κεντρική Μεσόγειο, αλλά και βελτιώνοντας ε, τις μυστικέ, μάλλον την ε, ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών και τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών αυτό αποτελεί τμήμα της απάντησής μας, της ανταπόκρισής μας στις προκλήσεις αυτές. Και θα συζητήσουμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε και στη συνάντηση στις 25 Μαΐου. Ο κύριος Επιτίδιος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ και την Ελλάδα και την Τουρκία. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ. Τους ε, εκτιμούμε και τους δύο και συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και έχουν καταδείξει ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί, να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένε προκλήσει, όπω για παράδειγμα τον τρόπο που συνεργάζονται στο Αιγαίο. Ένα από του λόγου που πετύχαμε άλλωστε στο Αιγαίο είναι ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μέσω των συμμάχων του ΝΑΤΟ κατάφεραν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ασφαλώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσω να είμαι πιο συντομό από ό,τι ήμουν τώρα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτό τον πρώτο γύρο. Ε, θα δώσουμε άλλα 11 λεπτά για το δεύτερο γύρο. Θα δώσω το λόγο σε όσο το δυνατό περισσότερου ομιλητέ γίνεται και ε, θα απαντήσει μετά ο Γενικό Δαματέα. Ξεκινάμε ξανά με τι ομάδε. Ο κ. Νταζόν. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε Αρκή. Κύριε Γενική Γραμματεία, η σταθερότητα που επικρατεί ή δεν επικρατεί ε, κάνει σαφή το ρόλο του ΝΑΤΟ ως ε, συλλογικό όργανο άμυνας ε, και αποτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νότια πλευρά μας, αστάθεια, αποτυχημένα κράτη, τρομοκρατία, εκεί ποια θα μπορούσε να είναι η αποστολή του ΝΑΤΟ, με ποιες ε, χώρες σκοπεύετε να συνεργαστείτε. Και σε ό,τι αφορά την, τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, ε, πιστεύω παραδόξως ότι ο στρατιωτικό, η στρατιωτική πτυχή της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι πολύ περιορισμένη. Ε, Παρόλο που είμαι πολύ μιλικαριστής κατά τα άλλα αμφιβάλλω για την ε, δυνατότητα χρήσης ε, της στρατιωτικής ισχύω σε μεγάλο βαθμό στον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άγνο. Ο κ. Μποστινάρου, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η συνεισφορά του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια τη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι τεράστια αν αντικατάστατη πρέπει να το πούμε όσο πιο ηχηρά γίνεται. Οι χώρες μας κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάσουν τις θεωτικές τους δαπάνες στο τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ τους. Είναι περιορισμένη αλλά σημαντική συνεισφορά από μέρους μας. Δύο ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την περιοχή μου. Εγώ είμαι Ρουμάνος αν δεν με ξέρετε. Πρώτον, πώς αξιολογείται την κατάσταση ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα. Βλέπετε μια τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εκεί. Και δεύτερον, σχετικό. Η Συρία δημιουργεί κίνδυνο η Ρωσία να χτίσει μια πρόσβαση στην, στην ε, Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Για το ECR, Κύριε Γενικαρματέα, ε, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ επίκαιρο γιατί η επίκαιρη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Στρατού. Το ανέφερε και ο κ. Γιούνκερ πέρσι στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ε, αυτό θα ήταν απειλή ενδεχομένω για το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Γερμανία... Ε, ε, δαπανά κάτι λιγότερο από 2% του ΑΕΠ της, αλλά ε, σε κάθε περίπτωση υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μια σύγχυση, ε, αλληλεπικάλυψη κλπ. μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή το 70, αντιστοιχούν στο 70% δαπανών του, επιχειρησιακών δαπανών του ΝΑΤΟ. ε, το θέμα. Ε, δεν είναι βέβαια ε, να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους πόρους και τα ίδια χρήματα και να τα ονομάσουμε διαφορετικά. Εδώ πρόκειται για καινούριο στρατό. Ευχαριστώ για τους πράσινους, κυρία Χάρμς. Πολύ πρόσφατα ήμουν στη Τρούκλα, στη Λιθουανία, στρατηγείο του ΝΑΤΟ και συζητήσαμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσουν με τους στρατιώτες εκεί που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα ποια είναι τα προβλήματά μας με τον αριθμό των στρατιωτών, με τις ε, ικανότητες, τις δυνατότητες που έχουμε, τους πόρους κλπ. Ε, δεδομένης της ε, σημαντικής αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια. Ε, πού ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο, σε ποια ακριβώς σημεία πρέπει να επενδύσουμε. Ε, αυτό το σκέφτομαι και εγώ και μου το είπαν και επί τόπου οι στρατιωτικοί. Ευχαριστώ η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας και κ. Σάφολ. Διαπιστώνω ότι για την Γαλλία ε, βλέπετε ότι οι προοπτικές είναι πολύ θετικές ό,τι αφορά την ε, Το πρώτο κόμμα της Γαλλίας όμως, ε, που μπορεί και να κερδίσει, είναι ε, υπέρ της εξόδου του, της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ. Γιατί? Γιατί το ΝΑΤΟ πολύ συχνά αποσταθεροποιεί τις περιοχές, γιατί είμαστε υπέρ μιας πολυπολικής, ενός πολυπολικού κόσμου, ε, το, για να σας δώσω παράδειγμα του Ιράκ ό,τι αφορά την αποσταθεροποίηση που μπορεί να επιφέρει τη δράση του ΝΑΤΟ. Και επίσης να υπογραμμίσω και το ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έρθουν σε σύγκρουση με τη Ρωσία, αυτή η σύγκρουση θα γίνει στο πεδίο της Ευρώπης. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει ούτε στην επικράτεια της Ρωσίας, ούτε στην επικράτεια των ΗΠΑ, δεδομένου ότι είναι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις. Οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια Γαλλία ισχυρή σε ένα πολυπολικό κόσμο. Θέλουμε να κατακτήσουμε αυτή τη δυνατότητα που αυτή τη στιγμή έχει η Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία έχει το 50% του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δεν έχει τρομακτικές οικονομικές δυνατότητες. Έτσι, το 50% του ΑΕΠ της Γαλλίας παρόλα αυτά έχει μια εξαιρετικά ισχυρή αμυντική ικανότητα. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα μας οδηγήσει σε μια αλλαγή του ίδιου του ΝΑΤΟ. Αυτό το είχε φανταστεί ο στρατηγός Ντεκόλ. Ήταν πάντοτε ε, εταίρος και θα είμαστε και εμείς εταίροι πάντοτε, αλλά απαιτείται και μια βαθιά αλλαγή στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Merci. Τέσσερα λεπτά. ακόμα. Ε, κύριε Μανέσκου. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα που είστε εδώ μαζί μας. Μετά από πολύ καιρό, όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε θετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία ε, μόλις έφτασε το 2% όσο κάποιες άλλες χώρες, λίγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η τάση είναι θετική, ε, κάτι που σημαίνει ότι διαθέτουμε πλέον περισσότερους οικονομικούς πόρους και, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, υβριδικές απειλές και ε, απειλές του κυβερνοχώρου κυρίως. Ε, πιστεύετε ότι αυτοί οι νέοι πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν κυρίως σε αυτές τις απειλές αυτή τη στιγμή αφιερώνονται πιο πολύ σε παραδοσιακές συμβατικές, συμβατικούς εξοπλισμούς. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την καταπλήρωση των κυβερνόπυλων. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η όψη για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ε, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία, που οθούν την Τουρκία όλο και πιο μακριά από τι κοινέ μα αξίε, κοινέ αξίε μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα θέλαμε να δούμε την Τουρκία εκτός του ΝΑΤΟ ή ακόμα και κάτι χειρότερο. Δεν θα ήθελα στο μέλλον η Τουρκία να μην είναι μέλο του ΝΑΤΟ, η Μαύρη Θάλασσα να μην ειναι μελο του ρωσική λίμνη και να δημιουργηθεί ε, από τη Μαύρη Θάλασσα, από τις χώρε τη Κεντρική Ευρώπη μέχρι την Αφρική. Ε, Κυρία Γκόμες, ε, οι, οι επιχειρήσεις ε, ασφάλειας στη θάλασσα, στη Λιβύη, ποιο λόγο έχουν αν ποτέ δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα ε, της ε, μεταρρύθμισης ε, του στρατιωτικού στη Λιβύη. Ε, αυτές οι επιχειρήσεις είναι τελείως άχρηστες. Μετά για την Τουρκία. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία. Η χώρα μας ήταν δικτατορία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και το ΝΑΤΟ ούτε που ενδιαφερόταν. Το ούτε και τώρα θα μας ενδιαφέρει το θέμα του κατά πόσον η Τουρκία κινείται προς την κατεύθυνση της δικτατορίας. Ευχαριστώ. Κύριε Στέτινα, ένα λεπτό παρακαλώ, έτσι ώστε να μιλήσουν όλοι όσοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ για το λόγο. Είπατε ότι ε, θα καλωσορίζατε μια μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ε, πριν από δύο χρόνια ε, το ΝΑΤΟ είχε εκφράσει μια κάποια ζήλια. Βλέπω ότι πια έχει εξομαλυνθεί. Ε, αλλά σε αυτή την περίπτωση, η περίπτωση μεγαλύτερη αυτονομία, πώ θα μοιραζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ τα καθήκοντα. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, ε, αντιμετώπιση τη Ρωσία. Ευχαριστώ και ο Σβάγκελ. Ε, πρόσφατα στηρίξατε την καινούρια κυβέρνηση της Μακεδονίας, λέει ο μιλτής. Ε, και ε, στα Σκόπια η υποστήριξή σας ήταν πολύ καλοδεχούμενη. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τη Μακεδονία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Διότι είναι απολύτως παράλογο εξαιτία του αποκαλούμενου θέματος του ονόματος μια χώρα που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και αποτελεί ακρογωνία ολίθο της σταθερότητας στην περιοχή να μην μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Uh, Ευχαριστώ κύριο Σκέλα. Δύο ερωτήσεις. Η κοινή διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ Τι έχει γίνει συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη αυτή. Βεβαίως προσβλέπουμε σε επιπλέον συνεργασία όπως ε, ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα. Δεύτερη ερώτηση. Επτά ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν δυνατότητες σε ό,τι αφορά την άμυνα στο χώρο. Το ΝΑΤΟ έχει διακηρύξει ότι τους ενδιαφέρουν μόνο οι αμυντικές δυνατότητες πώς θα αναπτυχθεί το ζήτημα αυτό στο μέλλον. Θα ενδιαφερθεί το ΝΑΤΟ για να αναπτύξει επιθετικές ε, δραστηριότητες δυνατότητες στο κυβερνοχώρο. Παράλληλα με τις ε, επιχειρήσεις της χερσές και τις ναυτικές. Και πότε θα δούμε κοινέ ασκήσεις στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η κυρία Ζάφκο τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, θέλω να ρωτήσω κι εγώ μαζί με άλλους ε, συναδέλφους σε σχέση με τον διφορούμενο ρόλο της Τουρκίας, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι θα λέγατε, τι θα κάνατε σε περίπτωση, όπως για παράδειγμα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, το ΝΑΤΟ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουμε διαφορετικούς παίκτες στις χώρες αυτούς. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίζατε αυτό το ζήτημα της έλλειψης δημοκρατίας στην, στην Τουρκία σε αυτές τις χώρες όταν ζητούσατε να εφαρμόσουν την αρχή της δημοκρατίας και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα κακό παράδειγμα ίσως και το ΝΑΤΟ διαδραματίζει σημαντικό ηθικό ρόλο. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εκπαιδεύουν τον στρατό στην Βοσνία λαμβάνουν ενεργή δράση, ενεργό ρόλο. Πείτε μας λοιπόν τι θα, τι θα κάνετε δημοσίως. Οι τελευταίοι τρεις ομιλητές, ο κύριος Κούκαν, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε Γενική Γραμματέα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, μετά την σύνοδο της ε, Βαρσοβίας, πώς βλέπετε την συνεργασία και ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής. Συγχαρητήρια για την ένταξη του Μοντενέγκρο, του Μαυροβούνιου στην ε, οικογένεια και πώς θα εξασφαλίσουμε το ζήτημα της ε, ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί οι χώρες αυτές αποτελούν ένα κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Θα πρέπει να εκφράσουμε έμπρακτα την ανησυχία μας. Ο κύριος Φροντζουλίκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, Γενικέ Γραμματέα. Με ενοχλεί το γεγονός ότι επιθυμείτε να είναι πιο έντονη η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και χωρίς βεβαίως να διπλασιάζουν να μιμούνται τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, αλλά να είναι συμπληρωματικές. Όσο έχουμε κοινά μέλη 22 χώρες και στους δύο οργανισμούς και οι δύο οργανισμοί υπερμάχονται των ίδιων αξιών, δεν θεωρείτε ότι είναι ίσως η ώρα για τους δύο αυτούς οργανισμούς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, ούτω ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν επιχειρησιακές συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ για αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως σε τρία πεδία, σε ό,τι αφορά το διάστημα, σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιχειρήσεις μεταφοράς εξοπλισμού και στρατευμάτων. Αυτά είναι εξαιρετικά παραδείγματα για τους κατοίκους του δυτικού κόσμου, για τους πολίτες του δυτικού κόσμου έμπρακτες αποδείξεις ότι υπεραμείνεστε των ιδίων αξιών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τελευταίος ε, παίρνει το λόγο ο Πέτερλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρκετοί συνάδελφοι ρώτησαν ερωτήσεις που αφορούν σε ειδικέ περιπτώσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τις δικές σας σκέψεις σε ό,τι αφορά την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, 26 άτομα πήραν το λόγο. Γενικέ Γραμματέα, τώρα εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε την πρόκληση του να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις όσο πιο διεξοδικά και όσο πιο σύντομα. Και αν δεν είχατε αρκετέ ερωτήσει, μια ερώτηση και από μένα. Η Αλβανία είναι μέλο του ΝΑΤΟ και περνάει μια περίοδο πολιτικής κρίσης. Υπάρχουν σχόλια από πλευρά σα, από πλευράς ΝΑΤΟ για την κατάσταση στην Αλβανία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω τώρα είναι να θίξω κάποια από τα ζητήματα που θίξατε και εσείς οι ίδιες ερωτήσεις σας. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν ονομαστικά στον, ε, στον καθέναν από εσά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από την Ρουμανία. Η Ρουμανία κάνει πρόοδους, διότι δήλωσε ότι θα φτάσει το 2% του στόχου που έχουμε ζητήσει. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν για τους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσουν το στόχο του 2%. Χαιρετίζω λοιπόν την προσπάθεια της Ρουμανίας. Ένα άλλο ζητούμενο ήταν οι κυβερνοαπειλές. Τι κάνουμε για τις κυβερνοαπειλές, οι υβριδικέ απειλέ, Κάνουμε πολλά. Προσπαθούμε όταν βρισκόμαστε σε υποεπίθεση στον κυβερνοχώρο έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αντιδράσουμε άμεσα, να αντιδράσουμε γρήγορα. Οι, οι εργασίες που κάνουμε στον κυβερνοχώρο έχουν να κάνουν με τις κυβερνοαπειλές, με τις υβριδικές απειλές. Έχουμε αυξήσει τις κυβερνητικές μας δίκαν ικανότητες, τα αμυντικά μας συστήματα, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να προστατεύσουμε τους δορυφόρους του ΝΑΤΟ. Έχουμε ε, οργανώσει ομάδες που μπορούν να αναπτυχθούν άμεσα σε διαφορετικά έθνη, σε διαφορετικές περιοχές που βρίσκονται υπό κυβερνοεπίθεση. Κάνουμε ασκήσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία του να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια κυβερνητική άμυνα απάντηση παράλληλα με τις χερσές και τις ναυτικές μας δυνάμεις. Και να βοηθήσουμε βεβαίως τα διάφορα κρατημέλη να κάνουν το ίδιο. Δεν ασχολούμαστε με την δυνατότητα επιθέσεων, αλλά βεβαίως αρκετοί συμμαχοί μας αναπτύσσουν τέτοιου τύπου δυνατότητες και θεωρώ ότι απάντησα σε αρκετά, αρκετές από τις ερωτήσεις σας θίγοντας αυτό το, το ζήτημα των κυβερνοαπειλών. Πώς ε, βλέπω τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μα, όπως σας είπα, σε σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν, έχουμε φτάσει σε ένα καινούριο επίπεδο συνεργασίας. Βεβαίως υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες, υπάρχουν προοπτικές, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά σε σχέση με το τι κάναμε προηγουμένως, έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Τον προηγούμενο μόλις χρόνο καταφέραμε να έχουμε δύο επίσημες συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τον κύβερνο χώρο και τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και αυτές είναι περισσότερες επίσημες συμφωνίες ε, που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια, μόλις ένα χρόνο λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Αρκετοί από εσά έθιξαν το ζήτημα της Τουρκίας και κάποιοι από εσά δήλωσαν ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την Ευρώπη, είναι σημαντική για όλη την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου έναντι στην, ε, στη μάχη ενάντια της τρομοκρατίας έχουν βάσεις, χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ τουρκικές υποδομές στην ε, μάχη ενάντια στο ISIS και κάποιοι από εσά βεβαίως ανησυχείτε για την κατάσταση στον Ευξενοπόντο και για την δική μας απάντηση στην ιδιαίτερη ανάπτυξη των ρωσικών δυνάμεων. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη, είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ να έχει την Τουρκία ως παρόντα σύμμαχο που συμβάλλει στην σταθερότητα στο Νότο, σε ό,τι αφορά το Ιράκ και την Συρία, αλλά προσπαθώντας να αναχαιτήσει και μια όλο και πιο έντονα παρούσα Ρωσία. Και πάλι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου είναι πυρηνικές αξίες για τον ΝΑΤΟ. Έχω αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτές τις αξίες, σε πολλές πόλεις συμπεριλαμβανομένες και της Άγκυρα. Και βεβαίως πάντοτε ε, στεκόμαστε σταθεροί στις αξίες μας και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάμε πάντοτε. Επίσης αναφερθήκατε στη Λιβύη. Συμφωνώ Απολύτως. Νομίζω ήταν ο κύριος Γκόμες που μίλησε για την Λιβύα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι ανάγκη να έχουμε ασφαλ... Ε, θεσμούς ασφαλείας. Γιατί αν δεν υπάρχει η σωστή υποδομή, τότε ίσως συμβάλλουμε και εμεί οι ίδιοι στην ε, κατάσταση αυτή αστάθεια Είναι ανάγκη λοιπόν το αμυντικό μας σχέδιο να περιλαμβάνει αυτές τις ε, υποδομές ασφαλείας. Είναι ανάγκη να έχουμε κοινέ δράσεις, είναι ανάγκη να έχουμε υπηρεσίες πληροφόρηση. πληροφόρησης. Έχω μιλήσει με αρκετούς ειδικού για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε στις περιοχές αυτές να, να χτίσουμε τις αμυντικές αυτές υποδομές. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θα πρέπει να, το αντιμετωπίσουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, τέθηκε το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις ευθύνες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μπορώ μόνο να μιλήσω εκ μέρους του ΝΑΤΟ και τα μέλη του ΝΑΤΟ που τυχαίνει να είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτά τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, η συλλογική ασφάλεια είναι ο βασικός στόχος, η βασική ευθύνη του ΝΑΤΟ. Γιατί η δύναμη αυτής της ε, συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ είναι ακριβώς η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Μπορούμε να πούμε πολλά για τον Καναδά, για, την, ε, για τη ΣΥΠΑ, όμως οι χώρες αυτές δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα. Είναι απλά σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί μετά μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές και μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί σε όλα μας τα σχέδια και σε όλους τους τομείς που θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας. Και όπως ανέφερα, ιδίω όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταλήψει, ε, φύγει, με φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το ΝΑΤΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε 80% του, του αμυντικού προπολογισμού του ΝΑΤΟ δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προέρχεται από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αφορούν αποκλειστικά το ΝΑΤΟ, τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ. Επιστρέφω τώρα στο ερώτημα που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμμαχία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πολλά από τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουμε δεν έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤΟ. Έχει να κάνει με αστυνόμευση, έχει να κάνει με υπηρεσίες πληροφόρησης, έχει να κάνει με ιδεολογικές μάχες που πρέπει να δώσουμε. Τομείς, με άλλα λόγια, με τους οποίους το ΝΑΤΟ δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά όμως το ΝΑΤΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται στο περιθώριο. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που μάχονται αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν, δεν μπορεί κανείς να τους πει ότι ο ρόλος τους είναι περιθωριακός. Ο μοναδικός λόγος που βρισκόμαστε στο Αφγανιστάν, που είμαστε στο Αφγανιστάν, είναι για λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε το ίδιο το Αφγανιστάν από την τρομοκρατική απειλή. Αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και δεν μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολεμούν εκεί πέρα ότι διαδραμάτισαν έναν περιθωριακό ρόλο. Έχουν χτίσει έναν στρατό στο Αφγανιστάν. Μια αποτελεσματική αστυνομία που μπορούν τώρα να αναλάβουν αυτοί οι ίδιοι τις ευθύνες προστασίας της ίδιας της χώρας τους. Κάνουν σκληρή δουλειά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το ΝΑΤΟ βεβαίως βοηθάει επίσης στην ε, συμμαχία που μάχεται ενάντια στο ISIS προσφέρει αεροπλάνα και εκεί ο ρόλος του ΝΑΤΟ δεν είναι περιθωριακός στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επομένως, ναι, υπάρχουν πάμπολα εργαλεία και κάποια από αυτά δεν έχουν να κάνουν με το, με το ΝΑΤΟ. Παρόλα αυτά όμως, η στρατιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ παίζει πολύ, σημαντική, πολύ σημαντικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί πρόσφατα ήμουν στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη και μου είπαν πόσο σημαντικό είναι να σταθεροποιήσουμε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα απαραίτητα εργαλεία, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και το ΝΑΤΟ και πάλι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενό στρατού στη Βοσνία. Είμαστε ακόμη παρόντες στο Κόσοβο, διατηρούμε δυνάμεις εκεί. Και φυσικά μας ενδιαφέρει η κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι δημοκρατίε οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές για την εκλογή κυβέρνησης. Και βεβαίως παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Αλβανία με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να επιληθούν. Η Αλβανία είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αυτά πιστεύω είναι τουλάχιστον τα περισσότερα που ρωτήσατε. Μία ακόμη από την κυρία Χάρντς γιατί χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ. Είμαστε ιδιαίτερα συγκεκριμένοι στο ΝΑΤΟ. Και θέλουμε ο κάθε ξεχωριστό σύμμαχος να προσφέρει κάτι διαφορετικό, πολύ συγκεκριμένο. Σε γενικές γραμμές όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο εξοπλισμό. Κάτι το οποίο δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου. Μας ενδιέφερε περισσότερο οι αποστολές στο Αφγανιστάν ή στα Βαλκάνια. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε πιο γρήγοροι, να μετακινούμε τα στρατεύματά μας ταχύτερα. Χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση, αναγνωριστικές ε, δυνατότητες, δυνατότητες παρακολούθησης, τόσο ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε τις απειλές και χρειαζόμαστε κάτι πάρα πολύ απλό, περισσότερες ασκήσεις, ούτω ώστε να είμαστε σε το επίπεδο ετοιμότητας να είναι καλύτερο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και είναι ανάγκη να τις αναπτύξουμε γιατί ζούμε σε μια επικίνδυνη περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Secretary... Κύριε Γενική Γραμματέα, στο Ολτενμπερέκ, εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, επικοδομητική αυτή συζήτηση από την οποία προέκυψε εκ νέου η αξία και η ανάγκη διατήρηση στενών δεσμών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και προσβλέπω στην συνέχιση των, ε, της ανταλλαγής απόψεων στις επόμενες συνεδριάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. And we now leave our και τώρα να αφήσουμε τους συναδελφούς της Επιτροπής, της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας να συνεχίσουν. Η κυρία Φωτίγκα. Σας παρακαλώ συναδελφοί της Υποεπιτροπής. Παραμείνετε στην αίθουσα και περιμένετε λίγο να χαιρετήσουμε τον